Πρόεδρος κυρία Βόλης. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μάρτιν, μετά την κυρία Ντόιλ, αλλά παρακαλώ να μην γίνει συζήτηση κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Μάρτιν, Hans Peter Μάρτιν. Την τελευταία φορά, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, όπως στην τελευταία πανηγυρική συνεδρίαση, ενδιαφερόταν ο πρόεδρο ιδιαίτερα για τη συνθήκη τη Λισαβόνα και παρενέβη όταν εκφράστηκαν άλλε απόψει. Σήμερα που έρχεται ο πρόεδρος μιας κυρίαρχη Δημοκρατία και λαμβάνει το λόγο και εκφράζει τι απόψει του και γίνονται μαζικέ διαμαρτυρίε από την πλευρά τη σοσιαλιστική ομάδα. Ο πρόεδρο δεν παρεμβαίνει για να τους, να τους ανακαλέσει την τάξη. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι δημοκρατία. Κυρία Ντόιλ, παρακαλώ. Μετά ο κύριος Μάρτιν Σούλτς. Κυρία Πρόεδρε, ένα διαδικαστικό σας παρακαλώ. Ναι, αν μου επιτρέψει ο πρόεδρος, θέλω να μιλήσω. Κατά τη γνώμη μου, μειώνει σοβαρά την αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου και του Τσέχου Πρόεδρου τότε επί τη ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης του πρόεδρου Κλάους υπονομεύεται επιτρέποντας να χρησιμοποιηθεί ευκαιρία για να μοιραστεί υλικό να επηρεάσουν την διαδικασία κύρωση τη ηθίκη τη Λισαβόνα. Διότι, κυρία Πρόεδρε, αν συμφωνεί αυτό με τον κανονισμό και περιμένω να αποφανθείτε, αν συμφωνεί, λέω, με τον κανονισμό, το λογικό συμπέρασμα θα ήταν μια συνταγή για χάο στου διαδρόμου. Καθένα που έχει το επιχείρημα το Α ή το Β να γεμίζει του διαδρόμου με άτομα που επιθετικά θα προωθούν τις απόψεις. Παρακαλώ διασφαλίστε ότι το Προεδρείο δεν θα επιτρέψει να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ κύριε Ντόελ. Κύριε Σούλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φωνάξτε μετά όταν θα ακούσετε ποτέ θα πω. Κυρία Πρόεδρε, μόλις ζήτησε το λόγο ένας συνάδελφος. Θα θυμίσω άλλα πράγματα. Όταν ο Πρωθυπουργός κ. Σόκρατες κατά τη διάρκεια της επίσημης υπογραφής του χάρτη των θεμελιών δικαιωμάτων επιθυμούσε να ομιλήσει δεν του επιτράπηκε εν τέλει διότι γίνονταν φωνασκίες και διαμαρτυρίες. Ο κύριος, Χάβελ, ο κύριος Κλάους μπόρεσε να μιλήσει. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δικών μας διαμαρτυριών και εκείνων. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Φομβόγκαου για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας και Άμυνας. Τροπολογία 10 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Για διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ξεχωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 11. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Όχι. Παράγραφος 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Δύο τροπολογίες. Πρώτη τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αν επιμένετε θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία νέα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 20 έχουμε δύο τροπολογίες. Τροπολογία 2, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Αν εγκριθεί, θα μετατοπιστεί σε άλλο σημείο του κειμένου. Μετά την παράγραφο 12. Αυτό προτείνει ο εισηγητής. Υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτή τη μετάθεση. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε τροπολογία 18. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 18. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Σαφέστατα. Παράγραφος 27. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 37. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Με Συγγνώμη, τροπολογία 15 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 15 στην παράγραφο 41. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. απορρίπτετε Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Για διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε ξεχωριστά τρεις παραγράφους. Πρώτα την 53. Παράγραφος 53. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ολόκληρο το σχέδιο ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. Το σχέδιο ψηφίσματος εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Επόμενο σημείο είναι η ψηφοφορία της έκθεσης Βατάνεν για το ρόλο του ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας. Το λόγο έχει ο εισηγητής Άρη Βατάναν για μια σύντομη δήλωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη που σας καθυστερήσω λίγο το μεσημεριανό φαγητό, αλλά μία φορά το κάνουμε κάθε 10 χρόνια. Ελπίζω λοιπόν να μην με παρεξηγήσετε. Ως ε, Φιλανδός Πρωθυπουργός Είχαμε έναν ε, Φιλανδό βουλευτή, ο οποίο το μόνο που είπε σα παρακαλώ κλείστε το παράθυρο». Μόνο αυτό η ευκαιρία του δόθηκε. Δεν ήθελα να πω δύο λόγια για το πακέτο αυτό. Ιδιαίτερα σε σχέση με τον Φοβάγκο και τον κύριο Σάρις Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για την οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή που την αυτοεπιβάλαμε και λέμε ότι δεν θέλουμε να επαναληφθούν τέτοιου είδου κρίσει. Ποιο είναι όμω ο λόγο ύπαρξη τη Ένωση να αποτρέπει πολέμους και ανθρώπινες κρίσεις. Αυτές οι κρίσεις δεν έρχονται ξαφνικά, δεν μας πέφτουν ορανοκατέβατα. Είναι δυνατόν να επαναληφθούν μόνο αν συνεργαστούμε. Θα το αποφύγουμε και σας θυμίζω η ειρήνη, συνάδελφοι παρακαλώ, η ειρήνη δεν είναι μονοπόλιο μιας μερίδας του κοινοβουλίου. Η ειρήνη ανήκει σε όλους. Η οικοδόμηση της ειρήνης είναι κοινός στόχος άνευ όρων. Είναι κάτι που δεν υπόκεινται σε όρους. Πρέπει να είναι κανείς ιδεαλιστής στη ζωή, να κοιτάει μακριά. Όταν τρέχεις μέσα σε ένα δάσος δεν κοιτάς μπροστά στα πόδια σου, κοιτάς μακριά να δεις πού θα πας, κοιτάς μακριά. Και έτσι πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε ομά ειλικρινείς και να θυμάμαστε γιατί έγινε η Ένωση. Για να Οικοδομήσε την ειρήνη. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, αυτό που θέλω να πω αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να σεβαστούμε την κληρονομιά του κυρίου Μονέ και των ιδρυτών της Ένωσης, ας ανήκουμε σε ένα κόμμα, το κόμμα που δημιουργεί ειρήνη. Το παράθυρο παραμένει ανοιχτό. Σας ευχαριστούμε κύριε Βατάνα Εδώ είναι ορθά ανοιχτά όλα τα παράθυρα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 25, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26, ονομαστική ψηφοφορία η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. εγκρίνατε. Τροπολογία 11. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 11. Ψήφισατε όλοι. Τέλος. εγκρίνατε. Τροπολογία 27 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 27. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19, συγγνώμη, παράγραφο 19, ποιο είναι υπέρ, ξεχωριστή ψηφοφορία, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 22, ψηφοφορία κατά τμήματα. Δύο είναι τα τμήματα. Ψηφίζουμε ονομαστικά το πρώτο τμήμα μόνο. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ο κύριος Βατάναν θέλει να προτείνει προφορική τροπολογία για την παράγραφο 29. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη που σας καθυστερώ και πάλι, απλώς θέλω να διαγράψουμε μία φράση για το Γενικό Επιτελείο υπογραμμίζει ότι το προτινόμενο επιχειρησιακό στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παρέχει τη λύση στο πρόβλημα. Αυτή τη φράση θέλω να διαγράψουμε. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Με την αλλαγή αυτή ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 20, ε, τροπολογία 22 για διαγραφή ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 15 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 4 καταπίπτει. Τροπολογία 24 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 24. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 και 23 που είναι ταυτόσιμες με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Έχουμε και μια προφορική τροπολογία του κυρίου Λαντσμπέργκης. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω δύο προφορικές τροπολογίες για την παράγραφο αυτή. Η πρώτη αφορά μια πολύ μικρή αντικατάσταση για τις ε, ανησυχίες μας. Ανθρώπινα δικαιώματα, και κράτος δικαίου θα πρέπει να προηγούνται ε, και όχι να έπονται στον κατάλογο, να είναι το τελευταίο σημείο. Και μετά την ψηφοφορία, ελπίζω να γίνει δεκτή αυτή η προφορική τροπολογία, θα σας παρουσιάσω τη δεύτερη. Ναι, αλλά είναι και την ίδια παράγραφο και οι δύο προφορικές τροπολογίες, οπότε καλύτερα να τις παρουσιάσετε μαζί. Μπορείτε να μας περιγράψετε και τη δεύτερη προφορική τροπολογία. Α, θα τις ψηφίσω μαζί. Η δεύτερη προφορική τροπολογία αφορά το δεύτερο τμήμα της παραγράφου. Τη Ρωσία ως δημοκρατία σε ένα προσδιορίστο μέλλον. γιατί υπάρχουν διάφορα, διάφορες έννοιες για το τι θα πει η δημοκρατία. Καλό θα ήταν να είμαστε πιο σχολαστικοί. Προτείνω λοιπόν μετά τον όρο δημοκρατία να προσθέσουμε το εξής. Και αρνείται τη στρατιωτική απειλή ως μέσο πολιτικής πίεσης προς τους γείτονες. Γιατί δεν είμαστε υπέρ τέτοιων πολιτικών, γι' αυτό και θα πρέπει να υπερψηφίσουμε την τροπολογία. Καλώ Για την πρώτη προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Για τη δεύτερη προφορική τροπολογία υπάρχουν ενστάσει. Ούτε. Ψηφίσουμε την τροπολογία 17 σε δύο τμήματα, όπως έχει τροποποιηθεί. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος της τροπολογίας 17, κατά, αποχές, εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Θεωρώντας 5, ονομαστική ψηφοφορία, η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη α, τροπολογία 7, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 για διαγραφή της αιτιολογικής σκέψης ε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη είναι ξεχωριστή ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 28 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ε, ψηφοφορία για την τροπολογία 28. Ψηφίσατε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 18. Ψηφίσατε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία για την τροπολογία 29. Ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 19. Ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το σχέδιο ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Βατάναν. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση Πασκογίνων Πολιτάνων για τη διαδικασία τη Βαρκελόνη Ένωση για τη Μεσόγειο. Ψηφίσουμε το ψήφισμα. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Υπέρ. Κατά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 κατά αποχές απορρίβεται. Τώρα το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. Έκθεση Σιμάνσκι. Ανεφιόρηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας το ψήφισμα. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπερφών 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Το επόμενο η έκθεση κ. Μπέρμαν, χρηματοδότηση δράσεων πλήν της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μπέρμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναπευθεί η έκθεση αυτή στην Επιτροπή με βάση το άρθρο 161, διότι το δημοκρατικά εκλεγμένο Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να καλυφθούν ορισμένε ήπιε μορφέ συνεργασία με τις Ένωση και ανεψόμενων χωρών τέτοιε δράσει, αλλά δεν είναι για την ελάφρυνση τη φτώχεια, διάφορε ανταλλαγέ προγραμμάτων με πανεπιστήμια Γι' αυτό δεν αναφέρεται αυτού του είδου η συνεργασία. Δεν προβλέπεται. Μερικά κράτη-μέλη επιμένουν χρησιμοποιηθεί μια νομική βάση που να μα οδηγήσει σε χρηματοδότηση αυτών των δράσεων με τον προπολογισμό ανάπτυξη. Αυτό ακριβώ θέλουμε να αποφύγουμε με την έκθεση αυτή. Δεν συμφωνήσαμε. Αν εγκριθεί η τροπολογία 1, η έκθεση αυτή θα είναι τελείω ανακόλουθη και αντίθετη με τα συμφέροντα των πιο φτωχών του πλανήτη. Γι' αυτό καλύτερα να επιστρέψει η έκθεση αυτή στην Επιτροπή Ανάπτυξη για να υπάρξει συμφωνία για την νομική βάση και να το υποστηρίξει σαφή πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, θέλει κανεί να μιλήσει υπέρ ή κατά τη πρόταση. Ο κύριο Γκάλερ, κατά νομίζω. Όντω, κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Όντω υπάρχουν διαφορέ απόψεων η άποψη της Επιτροπής Αναπτύξεως είναι αντίθετη με αυτήν της Επιτροπής Εξωτερικών, αυτήν της ε, Νομικής Επιτροπής, αντίκειται ακόμα στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και κατά της νομολογίας ε, του Δικαστηρίου, κατά ε, των, θέσεων Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό επιμένουμε στην νομική βάση όπως αυτή προκύπτει από την τροπολογία. Παρακαλώ λοιπόν να απορριφθεί η πρόταση εκ νέου παραπομπής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Επί της ουσίας δεν διαφωνούμε. Μόνο σε ό,τι αφορά την νομική βάση υπάρχουν απόψεις, ε, διαφορές απόψεων μάλλον, που δεν πρόκειται να απαλληφθούν ούτε και με την εκ νέου παραπομπή. Άλλος κανείς επιθυμεί να λάβει το λόγο υπέρ της απόψεως του εισηγητού. Η κυρία Γκόμες. Υποστηρίζω τον εισηγητή. Μετά από την συζήτηση που έγινε χθε εδώ, με συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ ότι όντως χρειάζεται περισσότερη συζήτηση και χρειάζεται αναζήτηση της σωστής νομικής βάσης για τις δράσεις αυτές, οι οποίες δεν είναι απλώς και μόνο ανάπτυξη, αλλά είναι αναπτυξιακή συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες. Και γι' αυτό δεν εμπίπτουν μεταξύ των άλλων μηχανισμών και πάντως όχι μέσα στο παρόν DCI. Και είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν τα χρήματα τα οποία είναι, προορίζονται για το DCI να είναι εξασφαλισμένο να θα χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτά. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο διαβουλεύσεων. Η πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε τώρα σχετικά με το εάν θα αναβληθεί ή όχι η ψηφοφορία και θα παραπεμφθεί εκ νέου στην Επιτροπή ε, το θέμα. Παρακαλώ ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. το επόμενο θέμα είναι για την έκθεση της κυρία Ντάλλα οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσία εκδόσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουμε το ψήφισμα. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τροπολογία παραθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία έναρξη ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας Και περάσουμε στην επεξήγηση ψήφου. Ο κύριο Σάμπερ πρώτο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εξηγήσω